Ε, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω. Ε, καλωσορίζω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μπούτικοφα και να περάσουμε στο θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά την Ουκρανία. Τη τελευταία εβδομάδα είχαμε την επικύρωση και θα ήταν καλό να πάρουμε περισσότερες εξηγήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί. Θα μπορούσα να αναφέρω και τη δική μου άποψη από αυτού. Έχουν υπάρξει σημαντικοί νόμοι, για παράδειγμα το ειδικό καθεστώς για την περιοχή Ντανιέτς και Λουγκάνσκ, ο νόμος ε, περί αμνηστίας και ο νόμος για το lustration. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς. Νομίζω πως ε, είναι σημαντικό να δούμε ε, τι περαιτέρω εξελίξεις θα έχουμε. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι 7 θα πάνε ε, ε, στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου. Θεωρώ πως είναι υπερβολικά μικρός αυτός ο αριθμός. Θα επιχειρήσουμε να ε, αυξήσουμε τον αριθμό. Έχω όμως και μία παράκληση. Να συζητηθεί στις πολιτικές ομάδες. Θα είχε έννοια. Ακριβώς πριν από τις εκλογές, πολλοί συνάδελφοι να πάνε στην Ουκρανία και μάλιστα όχι στο Κίεβο, να πάνε για να δείξουμε ακριβώς την παρουσία μας στο Χάρκοβο, στην ε, ε, Οδυσσό, να δείξουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι παρόν. Όλοι πηγαίνουν ε, στο Κίεβο. Όλες οι αντιπροσωπείες δεν εξυπηρετεί και ιδιαίτερα να συναντώμεθα μόνο με την κυβέρνηση. Τέτοιες αποστολές Ε, θα είχε έννοια. Θα είχε έννοια λοιπόν να πάμε και αλλού. Παρακαλώ λοιπόν να σκεφτούμε ποιοι θα μπορούσαν από ποια ομάδα πριν από τις εκλογές για να δείξουμε ακριβώς την παρουσία μας. Θα παρακαλούσα τώρα να μας παρουσιάσει ο Γκούνα Βίγκαντ το θέμα, πώς έχει η κατάσταση Ο κύριος Βίγκαντ είναι ο αρμόδιος και θα μας εξηγήσει πώς έχει κατάσταση στην Ουκρανία. Πού είναι ο κύριος Βίγκαντ? Ω, βλέπω ότι έχετε κάτσει πολύ μακριά. Θα σας παρακαλούσα να μας παρουσιάσετε την κατάσταση. Παρακαλώ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ε, πολύ ευγενική παρουσίαση. Να σας παρουσιάσω σύντομα τρία σημεία. Το πρώτο είναι εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Το δεύτερο είναι οι πολιτικές εξελίξεις μετά την έγκριση διαφόρων νόμων και τι περιμένουμε. Και τρίτον, τα περαιτέρω βήματα μετά την σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη Τρίτη στο Στρασβούργο. Πρώτον, όσον αφορά τα έγγραφα του Μίνσκ. Είχαμε το πρωτόκολλο των 12 ε, σημείων της 5ης ε, Σεπτεμβρίου για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και την ε, πολύ πιο αναλυτική την πιο αναλυτική εξήγηση του τι καθεστώς θα έχει η κατάπαυση του πυρός. Η ομάδα επαφής συμφώνησε και αυτά μας δίνουν ελπίδες ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση σε σχέση με την ένταση του Αυγούστου και ότι θα γίνουν περαιτέρω βήματα για μια βιώσιμη πολιτική λύση για τη σύγκρουση και για μία μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός. Μετά την ε, κατάπαυση του πυρός, το επίπεδο βίας στην περιοχή έχει μειωθεί. Και παρά το ότι οι πλευρές λένε ότι η κατάπαυση του πυρός ε, ισχύει, ε, αναφέρονται ακόμη επεισόδια βομβαρδισμών και πυροβολισμών στην περιοχή του αεροδρομίου του Ντανιέτσκ και μεταξύ Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ, η έγκριση του νόμου περί αμνηστίας. <clears throat> και, λοιπόν, η έγκριση των ε, ε, νόμων για την αμνηστία και για τη διακυβέρνηση των περιοχών και αυτό το πρωτόκολλο της 5ης Σεπτεμβρίου είναι ε, θετικά βήματα. Θα σας εξηγήσω αν θέλετε αργότερα τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η προσωρινή κυβέρνηση που σε μεγάλο βαθμό, η προσωρινή διακυβέρνηση που σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί τα αιτήματα των αποσχεστικών τάσεων και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι μια απόδειξη ότι θέλουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά το πρωτόκολλο παρά το ότι ήταν ε, πολύ δύσκολο βήμα για αυτούς και είναι πρωτοβουλία του Προέδρου Ποροσέγκο που προσπαθεί με διάφορα βήματα να δημιουργήσει μια, μια, βιώσιμη πολιτική λύση. Αλλά ο νόμος αυτός για την προσωρινή ε, τοπική αυτοδιοίκηση ε, θα ισχύσει για ε, το πολύ τρία χρόνια. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εντός της Ουκρανίας και υποθέτω ότι θα υπάρξουν έντονες συζητήσεις κατά την προεκλογική εκστρατεία της επόμενης εβδομάδας. Ελπίζουμε ότι η Ρωσία και οι αποσχετικές τάσεις θα δείξουν και αυτοί ε, θετική στάση θα ανταποκριθούν εφαρμόζοντας διάφορα σημεία της ε, συμφωνίας. Το πιο σημαντικό είναι η αποχώρηση των παρανόμων και ξένων ενόπλων δυνάμεων, του στρατηγικού εξοπλισμού, των μαχητών και των μισθοφόρων από την επικράτεια της Ουκρανίας, καθώς και μια μόνιμη επιτήρηση των συνόρων ε, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από παρατηρητές του. Όπως θα ξέρετε, στην στο πρωτόκολλο της 5ης Σεπτεμβρίου μιλούσαμε, ε, αναφέρονταν ο όρος παράνομες ε, ένοπλες δυνάμεις, ενώ στο πρωτόκολλο της 19ης Σεπτεμβρίου αναφέρεται και ο όρος ξένες ένοπλες δυνάμεις. Έτσι ελπίζουμε ότι θα αποσυρθούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτεια της Ουκρανίας υπό επιτήρηση και έλεγχο του ΟΑΣΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο του ΟΑΣΕ, και τις δυνατότητες ανταπόκρισης στην κρίση που έχουμε, διερευνούμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον ΟΑΣΕ, την ειδική αποστολή επιτήρησης του ΟΑΣΕ, να του στείλουμε ταχύτερα και εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται για να έχουν 500 επιτόπου που θα αναπτυχθούν ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η επιτηρήση που προβλέπουν τα δύο έγγραφα. Αυτή τη στιγμή κάθε εβδομάδα φτάνουν 25 επιπλέον παρατηρητές. Πρέπει λοιπόν να επιταχυνθεί αυτή η αποστολή προσωπικού και οι επιτηρητές βεβαίως πρέπει να είναι ειδικά καταρτισμένοι να μπορούν να επιτηρούν κατά του πυρός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως συμμετέχει και στηρίζει από πολιτική και διπλωματική πλευρά όπως συμφώνησαν μέσα Αυγούστου η Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης. Θα υποστηρίξουμε ενεργά οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται να υπάρξει μια νέα πολιτική πορεία. Είχαμε την ad hoc ε, προεδρική συνάντηση στις 26 Αυγούστου με συμμετοχή της ε, Άστον και των Επιτρόπων De και Oettinger. Στην Ολομέλεια αυτή δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την διμερή συνάντηση Ποροσέγκο-Πούτιν και έκτοτε έχουν γίνει πολλές διμερείς επαφές μεταξύ των δύο Προέδρων, οι οποίες βοήθησαν στο πρωτόκολλο του Μίνσκ και το καθεστώς για την κατάπαυση που αποφασίστηκε μετά. Η στήριξη στα πλαίσια της ε, δραστηριότητας της ομάδας επαφής και του ΑΣΕ και σε άλλα επίπεδα υψηλού επίπεδου θα ενταθεί ακόμη περισσότερο από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τι ε, αρμόδιε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, η διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων εντό τη Ουκρανία. Είναι αυτό ο χωρί αποκλεισμού ε, κοινωνικό διάλογο που ξεκίνησε πριν από τι προεδρικέ εκλογέ. Αυτό ήταν πάντα τμήμα τη συνολική πορεία μεταρρυθμίσεων για να υπάρξει μια μόνιμη πολιτική επίλυση τη κρίση είναι κλειδί για να υπάρξουν απαντήσεις ε, για θέματα συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και αυτοκέντρωσης στη χώρα. Αυτό ήδη αναφέρθηκε στο κοινό, στην κοινή δήλωση του Απριλίου της Γενέβης, όπου συμμετείχε και η Ένωση και τις τρογγυλές τράπεζες που έγιναν μετά. Γράφουμε τόσο σύντομα την ιστορία στην Ουκρανία που τα έγραφα αυτά συχνά πάνε στο καλάθι. Αλλά είχαμε το μνημόνιο για ειρήνη και ομόνια που εγκρίθηκε στις 21 Μαΐου. Μετά τις προεδρικές εκλογές η διαδικασία επιβραδύνθηκε. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι είχαν ε, ήδη προκηρυχθεί πρόορες κοινοβουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στις 26 Οκτωβρίου. Και αυτό είχε επίπτωση βέβαια και βεβαίω και ιδιαίτερα επισφαλής κατάσταση ασφαλείας παίξει ρόλο. Η προεκλογική εκστρατεία βεβαίω είναι τώρα σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά δεν είναι το πιο κατάλληλο περιβάλλον για δημιουργία ε, συνένεσης. Αλλά, τονίζω, χρειαζόμαστε την ενίσχυσή σας στις πολιτικές επαφέ σα με πολλούς Ουκρανούς εταίρου. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ε, συνταγματικέ, αποκέντρωση, της δικαστικής εξουσίας και του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων. Όλα αυτά έχουν καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ είναι τμήμα των προτεραιοτήτων μεταρρυθμίσεων με βάση το θεματολόγιο της Συμφωνίας ε, Σύνδεσης και της, ε, του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για Μεταρρύθμιση. Εάν λοιπόν επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες, θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες προσδοκίες ε, της κοινωνίας των πολιτών. Και ελπίζουμε η προεκλογική διαδικασία να οδηγήσει σε μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανική Βουλή. Τι ράντα μακροπρόθεσμα πρέπει οι διαδικασίες αυτές να συνεχιστούν και μετά τις εκλογές. Πρέπει να στηρίξουμε πλήρως αυτές τις διαδικασίες και το κάνουμε καθημερινά τώρα που έχουμε και την ομάδα στήριξης της Ουκρανίας που είναι πλήρως λειτουργική. Προσπαθούμε να του ενθαρρύνουμε. Αυτό ο χωρίς αποκλεισμού ε, κοινωνικός διάλογος είναι στοιχείο του πρωτοκόλλου του Μίνσκ τη 5 η Ανάτου. Τονίζω ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν και δημοκρατικά νομιμοποιημένοι εκπρόσωποι του Ντανιέτ και του Λουγκάνσκ που να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε οι κοινοβουλευτικέ εκλογέ και μετά οι προώρε εκλογέ ε, τοπική αυτοδιοίκηση που θα γίνουν σε αυτά τα ομπλάστ να βοηθήσουν και να οδηγήσουν με πλήρη ε, επιτήρηση σε δίκαιες εκλογές. Τώρα, για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης. Η παράλληλη επικύρωση από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, Ναχόβνα Ράντα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Και αυτό μας βοήθησε για να προχωρήσουμε σε πολιτικές σχέσεις και οικονομική συνεργασία. Η συμφωνία αυτή, ελπίζουμε, να αρχίσει να εφαρμόζεται προσωρινά πρώτη ενδεκάτου μετά την ε, ε, ενημέρωση από τη Ράντα και την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός βέβαια από το κεφάλαιο 4 που αφορά το εμπόριο για το οποίο η προσωρινή εφαρμογή θα αναβληθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2016 μετά από τη συμφωνία που επετεύχθη στις 12 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ε, Υπουργών Λουκάευ Ρωσία, Κλίμκι ε, Ουκρανία και τον Επίτροπων αυτό σας τα εξήγησε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Ντεχούκτα στην Ολομέλεια. Η Ρωσία συμφώνησε σε αντάλλαγμα να συνεχίσει να εφαρμόζει το καθεστώς προτιμήσεων για τις εμπορικές σχέσεις. Και οι τρεις πλευρές συμφώνησαν ότι θα συνεχιστούν οι διαδικασίες διαβούλευσης που θα είναι τμήμα μια συνολικής επίλυσης για την επίτευξη ειρήνης, σεβόμενη βεβαίως ε, το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει για το μέλλον της και, για, και σεβόμενη βεβαίως και την ε, εδαφική ακαιρεότητα. Αυτό είναι ήδη μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ασύμετρης φιλευθεροποίησης, διότι δεν θα εφαρμόσουμε λοιπόν αυτό το τμήμα για το εμπόριο όπως είπα, αλλά παρόλα αυτά θα ζητήσουμε να επεκταθούν, δηλαδή να παραταθούν τα αυτόνομα μέτρα εμπορίου και θα αποστείλει η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο πρόταση εντό των ημερών. δυστυχώ η ρωσική πλευρά παρά το ότι δέχθηκε την δήλωση των τριών υπουργών ερμηνεύει με πολύ στενό τρόπο αυτά που ε, συμφωνήθηκαν και ο Υπουργό Μουλουκάιεφ έστειλε στον Επίτροπο Ντεχούκ και τον Υπουργό Κλίντ μία επιστολή όπου εξηγεί την ε, άποψή τους στις 9 Σεπτεμβρίου. Υπήρξαν κάποιες μονομερείς ενέργειες από πλευρά τη ρωσική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργό Μετβέντεφ υπέγραψε ένα διάταγμα που αναστέλει την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής για την Ουκρανία με βάση το παράρτημα 6 αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και είπε ότι θα συμφωνηθεί ε, ότι θα εφαρμοστεί αυτό το διάταγμα που δεν θα επιτρέπει το ελεύθερο εμπόριο εάν αρχίσει να εφαρμόζεται η Συμφωνία Σύνδεσης. σε αυτέ τι ε, αποφάσει της κυρίαρχε, οπότε θα ξεκαθαριστεί το τι γίνεται όσον αφορά το πώ θα ε, ανταποκριθεί η ρωσική ηγεσία. Σε σχέση λοιπόν με την Ουκρανική ηγεσία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, το παρακολουθούμε και την κατακλείδη τώρα θα υποβάλουμε όλα αυτά στο Συμβούλιο για να αλλάξει η απόφαση της 26 ης του Συμβουλίου και έτσι να καθυστερήσουμε ε, την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθερών Εμπορίου, αλλά εν όλα αυτά ε, θα σας τα και εσάς και το Συμβούλιο, ούτως ώστε να επεκτεθούν αυτά τα αυτόνομα μέτρα ε, που φτάνουμε το 2015 και οπότε και σε αυτό το διάστημα θα υποφερθούμε αυτή την οικονομική και τόσο να συνεχιστεί η διαδικασία διαβούλευσης και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες των Ρώσων και σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος εγώ σας ευχαριστώ πολύ Thank you very much, Mr. Chairman. Thank... Σας ευχαριστώ, ο κύριος Πλέγκοβιτς. Δεν μπορώ παρά να τονίσω το ότι το Κοινοβούλιο θα ήθελε να έχει μεγαλύτερη ε, ομάδα παρατηρητών για τις εκλογές του 26ου και είπαμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι που ανήκουν στην αντιπροσωπεία των σχέσεων με την, Ουγγαρία, ή με την ε, Ουκρανία θα ήθελαν να συμμετάσχουν οπότε και η ΑΦΕΤ θα απευθυνθεί στην διάσκεψη των Προέδρων, τόσο ώστε να διευρυνθεί η σύνθεση της ομάδας των παρατηρητών λόγω της σημασίας ε, του γεγονότος αυτού, των εκλογών δηλαδή στην, στην ε, Ουκρανία. Έχουμε δύο κεχηρίες, δύο καταπαύσεις. Πρώτα-πρώτα είχαμε μία που την ε, ασφάλεια μέσω των επαφών του Μίνσκ με τις τριμερείς επαφέ και αυτό ενισχύθηκε από τη συμφωνία της 19ης και είχαμε εδώ κάπως πιο ενδελεχείς ρυθμίσεις όσον αφορά τι εφαρμοστικές λεπτομέρειες της κατάψης του πυρός ε, και σε σχέση με τον ΟΑΣΕ ε, οπότε και τότε ε, είχαμε κάποιου παρατηρητές για να υποπτεύσουν την υλοποίηση της για γιατί πηγές πληροφορούν από τη Ρουμανία ε, παρά την διαχειρία μας είπαν είχαμε πάνω από 19 νεκρούς ε, επίσης και θύματα εν μέσω των αμάχων. Κατά αυτή την περίοδο δηλαδή το, η καινούργια διαχειρία ελπίζουμε ότι θα είναι ένας ε, προάγγελος ειρηνικών εκλογών. Τώρα επίσης είχαμε τη συμφωνία των Βεξελών του Ντεχίχτ και των Υπουργών από Ρωσία και Ουκρανία. Βασικά θέλαμε να μην ε, γίνουν περαιτέρω μέτρα οικονομικά κατά τους κανείς από την Μόσχα και επίσης ε, έχουμε και την χειρονομία της Αγωγικής Ένωσης για ε, αυτή την ενίσχυση μέσω της συμφωνίας που θα γίνει σε 40 μήνες οπότε είπαμε ότι αυτό είναι κάτι το αναγκαίο, είναι μια θαραλέα απόφαση από όλου τους εμπλεκομένους και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε μια πιο ε, νυφάλια αντιμετώπιση του τι θα γίνει ε, τον χειμώνα ο οποίο έρχεται και έτσι ελπίζουμε ότι οικονομικά θα ενισχυθεί η Ουκρανία. Τρίτο θέμα, κατά τη γνώμη μου, ε, είναι το πιο κρίσιμο και είναι η δική μας αρρωγή όσον αφορά την υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης, γιατί πολλοί εξημών έχουμε ε, ασχοληθεί ε, γιατί η χώρα μας ε, τελικά είχε τέτοια συμφωνίες και μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν για να έχουμε ένα σωρό μεταρρυθμίσεις σε κάθε πεδίο ε, οπότε και γι' αυτό και έχουμε την ε, ομάδα υποστήριξη της ε, Επιτροπής για αυτή την υλοποίηση, έχουμε την χρηματική ενίσχυση, αλλά από την άλλη μεριά να έχουμε μια ξεκάθαρη συνεργασία για διάφορα νόμους και νομοσχέδια και τελικά αυτό το πακέτο το οποίο εγκρίθηκε με αυτή την ταυτόχρονη έγκριση με την αμνηστία, με την συμφωνία σύνδεσης, με τι ρυθμίσει για Ντονιέ και Λουχάνσκ, Όλα αυτά τελικά ήταν πολιτική κίνηση πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι επικοδομητικό λιθαράκι ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, να εξασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα και κατά τις ε, διασκέψεις μας και τις επαφές να μην ξεχνάμε την Κρυμαία. Διότι, διότι και εκεί πρόκειται για αθέμητη παράνομη προσάρτηση και οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παραλαμβάνει ε, στο ψήφισμα μας τελευταίας εβδομάδας στο Στασβούργο αυτή τη θέση. Και θεωρώ ότι οι κοινωνικές εκλογές πρόκειται να δημιουργήσουν ένα νέο τοπίο πολιτικό στην ε, Ουκρανία, θα ενδυναμώσουν την δημοκρατική νομιμότητα σύμφωνα με τη θέληση του Ουκρανικού λαού που θέλει να έρθει στην Ευρώπη, να φτάσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ και το Κοινοβούλιο και η Γενικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες της πλειοψηφία του Ουκρανικού λαού για τους ε, επόμενους μήνες. Δεν περίμενα να είμαι ο πρώτος. Εν πάση περιπτώσει έχω μια σύντομη ερώτηση. Εκπλήσωμαι που αυτή η κατάρριψη τραγική του αεροσκάφους που συνέβη στην, σε ουκρανικό έδαφος δεν αναφέρθηκε καθόλου. Ούτε στα πλαίσια της πάυσης του πυρός, ούτε ούτε σε, σε σχέση με οτιδήποτε αναφέρθηκε σήμερα εδώ. Ξέρουμε ότι ήταν πάνω από 300 άνθρωποι, 370, οι οποίοι ήταν απολύτως αθώοι και έχασαν τη ζωή τους σε ένα δυστύχημα το, το οποίο τα αίτια ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί, δεν έχει επιληθεί. Ρωτώ λοιπόν, έχουν υπάρξει βήματα έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι για το τι έγινε. Επίσης, τι συμβαίνει με τις ορούς αυτών που βρίσκονται ακόμα επί τόπου. Τι συμβαίνει με τα συντριμμία του αεροσκάφους, τα οποία επίσης βρίσκονται ακόμα επί τόπου. Θα ήθελα να ακούσω μερικά πράγματα σχετικά με το ατύχημα αυτό. Ευχαριστώ. Uh, thank e Ευχαριστώ πολύ. Ε, Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να πω ότι ε, οπωσδήποτε η Ουκρανία σαν, ε, ε, σαν κράτος έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την εξωτερική της πολιτική με τον τρόπο τον οποίο θέλει να τον κάνει. Ε, ωστόσο, από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι παραβιάσεις ε, του κράτους δικαίου και επίσης υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι τα ε, αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία έδωσε η Ρωσία βρίσκονται, είναι η αιτία της κατάρρευσης του αεροπλάνου. Εν πάση περιπτώσει ξέρουμε επίσης ότι διαρκώς ε, ε, μέσω της βίαιης επιθετικής συμπεριφοράς η Ρωσία σαφώς παραβιάζει τις αρχές της χάρτας. Εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι κάθε φορά ο στρατός της Ουκρανίας προσπαθεί να αγωνιστεί κατά των ανταρτών και και κάθε φορά έχουμε παρέμβαση των ρωσικών στρατευμάτων. Αυτό που με απασχολεί και νομίζω ότι και ο πρόεδρος Χέλμαν Μπρόκ επίσης ε, συμφωνεί με την άποψη αυτή την έχει ήδη εκφράσει είναι ότι σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε είναι ότι υπάρχει μια ε, άποψη στους εμπειρογνώμονες και τους διπλωμάτες ε, στο Κίεβο ότι η παράνομη προσάρτηση της ε, Κρυμαίας δεν θα έχει δυνατότητα επιβίωσης εάν δεν δοθεί κάποιος χερσαίος διάδρομος και νομίζω, ότι με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουν στρατιωτικά να πιέσουν έτσι ώστε να ανοιχτεί αυτό, αυτός ο διάδρομος ε, που θα συνδέει με την Ρωσία και επομένως ε, οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν νέα προβλήματα, κυρίως μια και ο χειμώνα βρίσκεται πρώτων θυρών. Τι θα κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε περίπτωση κατά την οποία θα γίνει προσπάθεια ε, να διανοιχτεί αυτός ο διάδρομος για να υπάρχει η άμεση επαφή με την Κρυμαία και ποιες είναι οι προληπτικές κυρώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και επίσης τι δυνατότητες μπορούν να δοθούν στον Ουκρανικό στρατό έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Thank you, Chairman. <coughs> Colleagues, indeed we have to... Έχουμε την ταυτόχρονη κύρωση τη Συμφωνία Σύνδεση και τη Συμφωνία Ελευθερία Εμπορίου στο Κίεβο. Αυτό είναι γεγονό ιστορική σημασία και σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ παγκοσμίω φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι αυτό και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση και θα πρέπει να γίνουν όλα τα πράγματα από πλευρά πολιτικών χειρισμών σωστά. Χρειάζεται επομένω πολιτικό θάρρος πρώτα πρώτα από την Ουκρανική ηγεσία και από τα πολιτικά κόμματα και θα πρέπει και εκείνοι να οδηγήσουν την χώρα σε ένα διαφορετικό μέλλον. Πάντως ζήτησα το λόγο για να σας πω ότι είμαι λιγότερο θετικός και αισιόδοξο όσον αφορά το εξή. Αυτές τις συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας ούτως ώστε να επηρεάσει, να χειραγωγήσει ακόμα και τις διμερείς επαφές και διμερείς συμφωνίες Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσον αφορά επίσης την καθυστέρηση της εφαρμογής της συμφωνίας του εμπόριου, και αυτό είναι σημείο αδυναμίας, παρά το το προσέχουμε αλλιώ. Και επομένως, να, πόσο από ό,τι χαρακτηρίζεται η πολιτική μας για να μην ξεχνούμε ότι οι Ρώσοι οι Υπουργοί και ο ίδιος ο κύριος Πούτιν συνεχώς απαιτούν από τις Ουκρανικές ε, αρχές να παρατηθούν από τις περαιτέρω αλλαγές που χρειάζονται ούτω ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία που κυρώθηκε. Ενώ οι Ρώσοι συμφώνησαν, θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαν αυτό να το θεωρήσουν ότι είναι η πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι έτσι. Θέλουν να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία παρά αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις. Και εάν εμείς δεχθούμε ότι είναι κάτι το de facto αυτή η ανάμειξη της Ουκρανίας σε αυτές τις δημιουργίες μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τότε φανταστείτε τι έχει να μας βρει τους αμέσως πόμους μήνες ή και χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι εάν οι εξελίξεις στην Ουκρανία μας οδηγήσουν στο να παρακολουθήσουμε από κοντά τις εξέλιξεις για την υλοποίηση της συμφωνίας, ε, τότε αξίζει να έχουμε μια μόνιμη ομάδα εποπτείας εδώ στην ΑΦΕΤ. Και έτσι να μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε ημερήσια βάση τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Αλλά γιατί όχι και τις νομικές σε σχέση με αυτήν την συμφωνία. πολιτική μας ομάδα Θέλει επίσης να επαναλάβει το ότι είμαστε συνεπώς ε, υπέρ αυτής της ε, πολιτικής γυτνίασης με τις χώρες Πασαντολάς και επομένως θα πρέπει αυτή η ομάδα εποπτείας να συνεργαστεί με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Κομισιόν, να έχουμε τις αναγκαίες πληροφορίες, ούτως ώστε να μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα που πρέπει σε όλους εμπλεκομένους. Γενικώ είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η ΑΦΕΤ ασχολείται με τη συμφωνία αυτή. Και θα πρέπει τα πράγματα να ξεφύγουν του ελέγχου μας. Τα πράγματα πρέπει να πάρουν το δρόμο τους, το σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Gracias, Bueno, para nosotros nos sigue pareciendo un... Πρόεδρε, όλα αυτά που έγιναν στην Ουκρανία μας φαίνονται απαράδεκτα. Η ομάδα μου θεωρεί ότι έχουν, ε, έχει υπάρξει ένα πραξικόπημα με βάση την, ε, με, και τη συμμετοχή και να ζεστών και είμαστε κατά των κυρώσεων. Θεωρούμε επίσης ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά, ε, αν, θεωρούν, αν δούμε τι έγινε στη Γάζα. Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα οι αγρότες στη χώρα μου να μην μπορούν να εξάγουν γεωργικά προϊόντα και η Ρωσία βεβαίως αμέσως βρήκε ε, άλλους για να αγοράσει αυτά τα προϊόντα από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και δύσκολο λοιπόν θα επανακτήσουμε αυτή την αγορά. Η εμπορική συμφωνία και η συμφωνία σύνδεσης δεν νομίζουμε ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι σκόπιμο να συζητηθεί. Θεωρούμε ότι είναι απόλυτη παντομήμα και έλλειψη σεβασμού αυτό που έκανε ο Σούλτ στο Κοινοβούλιο. Και θα προσφύγουμε κατά αυτής διαδικασίας. Δεν έδωσε ούτε καν το λόγο στην ομάδα μας για διαδικαστικό θέμα. Θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τι γίνεται. Θα ε, παρακολουθήσουμε και στην Ουκρανία, θα πάμε. Ξέρουμε ότι τέθηκε σε παρανομία το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βεβαίως, ε, είμαστε υπέρ της ειρήνης. Θέλουμε να γίνουν διαπραγματεύσεις. Εγώ ε, θα ήθελα να ε, ε, μιλήσω για το ε, αεροπλάνο της Μαλαισίας που δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Και επίσης πάλι δύο μέτρα και δύο σταθμά γιατί να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ουκρανία σε σχέση με το Κωσυφοπέδιο για παράδειγμα και να προσέχουμε διότι αυτά τα οποία λέμε δεν είναι ελεγμένα. Χρειαζόμαστε μια ε, ευρωπαϊκή πολιτική χωρίς παρέμβαση των ΗΠΑ και για το μέλλον της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε καλή γειτονία με την Ρωσία, άρα πρέπει να επιχειρήσουμε να την επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σωστά προφέρατε το όνομά μου. Θα ήθελα να προειδοποιήσω την Επιτροπή μας λέγοντας ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι πολύ σύντομα μετά την Συμφωνία Σύνδεσης. Και τι λέμε, ευχολόγια, ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η προειδοποίηση. Πρώτα απ' όλα η κατάσταση ασφαλείας. Είμαστε στο έλεος ε, της Ρωσίας του Πούτιν. Η παρατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και άλλα 25 επιπλέον άτομα τη βδομάδα. Τίποτα δεν είναι αυτό για να μπορεί κανεί να παρακολουθεί μια συμφωνία κατάπαυση του πυρό. Χωρί τον ΟΣΑ, χωρί ο ΑΣΕ, συγγνώμη, να έχει πιο ουσιαστική παρουσία, πιο πολυάριθμη για να μπορεί να παρακολουθεί τα σύνορα αυτά, τα Ουκρανο-Ρωσικά σύνορα, δεν θα υπάρξει σχετικά σταθερή κατάσταση ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα συνεχιστεί το, πρόγραμμα, το πρόβλημα, συγγνώμη, οποιοδήποτε και αν είναι στην κυβέρνηση του Κιέβου. Τώρα εγώ δεν έχω καμία πανάκια να σας προτείνω, αλλά προειδοποιώ την Επιτροπή μας ότι αν δεν υπάρχει σωστή παρατήρηση και της εφαρμογής της αποκέντρωσης, δεν θα υπάρξει πολιτική λύση. Αυτά είναι τα δύο σημεία κλειδιά οποιασδήποτε πολιτικής λύσης τώρα για την οικονομία θα εφαρμοστεί η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μόνο το 2016 θα αρχίσει να εφαρμόζεται αλλά γενικά ανησυχούμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την κατάσταση πριν λήξει αυτή η θητεία γιατί οι συμφωνίες εμπορίου δεν έχουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα για την κοινωνία, για τους πολίτες επιτόπου Πρέπει λοιπόν ε, τα επόμενα χρόνια να επιτηρούμε την εφαρμογή της. Εν κατακλείδη. Βεβαίω, συμφωνώ με τον Πρόεδρο, περισσότεροι εκλογικοί παρατηρητέ. Τι, με 7 άτομα, είναι γελίο. Με 7 άτομα θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει σε ε, κοινοβουλευτικέ εκλογέ στην ανατολική πλευρά τη χώρα. Και εκεί είναι το τι θα γίνει το σημαντικό, όχι τι θα γίνει στο Κίεβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα τα διπλά μέτρα και σταθμά. Ε, ε, μιλάμε για αποκέντρωση στην Ουκρανία και ταυτοχρόνως λέμε ότι υπάρχει ανάγκη ε, σεβασμού των αρχών της αυτονομίας, ας πούμε, της ε, Ουκρανίας. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα δούμε τι θα γίνει όταν θα αποφασίσουν, όταν αποφασίσουν οι Ουκρανοί να προσεγγίσουν την Ευρώπη. Και βεβαίως διάφορα μέτρα τα οποία προτείνονται ε, στην ουσία σημαίνουν ότι δεν σεβόμαστε την ε, ε, εθνική κυριαρχία της, της Ουκρανίας. Όσον αφορά τώρα το monitoring group, ναι, πράγματι θα πρέπει να διευρυνθεί, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει, εάν και εφόσον διευρυνθεί, να συμπεριλάβει και τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες εκφράζονται και για και από την Ουκρανία και νομίζω ότι αυτό θα είναι τόσο το, αυτό είναι είναι το σημαντικό. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ε, αμοιβαιότητα σε περίπτωση που υπάρξει διεύρυνση αυτού του monitoring Δεν κατάλαβα πολύ καλά ε, ποια είναι η διασύνδεση της επιχειρηματολογίας σας ανάμεσα στην αποκέντρωση και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας. Μου διέφυγε λίγο. Εγώ έλεγα ότι ε, θέλουμε να δώσουμε, ε, ότι πρέπει να δούμε πιο μακροπρόθεσμα την ε, κατάσταση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να στηρίξουν το ενδεχόμενο να μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί αναφερόταν η επιχειρηματολογία μου. Εν πάση περιπτώσει είναι πολιτικό σημείο. Πρόεδρος, ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί. Εγώ θέλω να καταλάβω οι λογικοί που βρίσκονται πίσω από επιχειρήματα, τα οποία ενδεχομένως δεν είναι δικά μου ή δεν τα συμμερίζομαι, αλλά θέλω να τα καταλάβω. Υπάρχει ένα σαφής κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι κάθε χώρα έχει εθνική κυριαρχία όσον αφορά την εσωτερική της οργάνωση. Το αν θα έχουν επικέντρωση, αποκέντρωση ή οτιδήποτε άλλο είναι δικιά τους απόφαση. Η εσωτερική δομή της χώρας τους είναι ε, απόφαση η οποία αφορά την εθνική τους κυριαρχία και είναι δικό του θέμα, γι' αυτό μου διέφυγε η επιχειρηματολογία σας. Χωρί μικρόφωνο οι διερμηνείς δεν ακούν. Οι διερμηνείς εξακολουθούν να μην ακούν. Κοιτάξτε, ναι, καταλαβαίνω τι σημαίνει φεντεραλισμός, φεντεραλισμός ομοσπονδοκράτος και, από και, και αποκέντρωση. Διαφορετικά εννοούμε εμείς στη Γερμανία, διαφορετικά εσείς ε, στην Βρετανία. Εμείς ε, εδώ μιλάμε για αποκέντρωση. Ναι, ναι, βέβαια, εγώ τα βλέπω πάντα από τη Βρετανική σκοπιά. Ωραία, τώρα εμείς μιλάμε μεταξύ ε, κυριάρχων κρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς και όλοι συμφωνούμε ότι η Ουκρανία δικαιούται να διαμορφώσει τη δική της ιστορική πολιτική και να διαλέξει τους συμμάχους της, εκείνους που ευθυγραμμίζονται με τις επιθυμίες της, με το τι θέλει ο λαός της χώρας. Όμως, σας τονίζω ότι Βεβαίω και θέλουμε να πριτανεύσει η ειρήνη στη χώρα, όμω να συνειδητοποιήσουμε ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μα χρειάζεται αυθεντική πολιτική βούληση από όλε τι πλευρέ. Η Ρωσία δεν έχει τέτοιου είδου πρόθεση. Στρατηγικό τη στόχο είναι η Ουκρανία να μείνει στη σφαίρα επιρροή τη. Και αυτό να γίνει με κάθε μέσο. Και χρησιμοποιεί και χειρία για τον αυτό τον διάδρομο προς την ε, Κρυμαία και ακόμα παραπέρα ε, κατά μήκο των ακτών της, ε, του Ευξηνού Πόντου. Και επίσης αυτού του είδους το κομβόι, το ανθρωπιστικό, αυτό έδειξε ότι μετέφεραν τότε υλικά ραδιοπικοινωνίας, όπλα, κατασκόπους, πυρομαχικά με εκείνο το ανθρωπιστικό κομβόι. Και μας το λένε οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ότι ε, ακόμη δεν έχουν λάβει οι αυτονομιστές ε, αυτά τα υλικά ε, ραδιοεπικοινωνίας. Και επίσης, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, δεν πρόκειται να αποσύρει η Ουκρανία τις δυνάμεις της πίσω από την ουδέτερη ζώνη. Διότι ποτέ πραγματικά δεν εφαρμόστηκε η εγκεχηρία εκεί οι συνάδελφοι, ευρωβουλευτές, απευθύνομαι σε εσά. Καταλάβουμε όλοι ότι η Ουκρανία χρειάζεται στρατιωτική βοήθεια ούτω ώστε να μπορέσει να ισχυροποιήσει ε, τις δυνατότητες ε, εθνική άμυνα. Όπως κάθε κράτο μέλος ε, πρέπει να αποφασίσουμε κι εμείς το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ίσως μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον στρατό της χώρας. Μπορούμε να δώσουμε κάποιο είδου όπλα, ε, τόσο πάντων στρατιωτικό υλικό, είτε όπλα είτε άλλο υλικό. Και έχουμε και την επιστολή ολουκέφ ότι δηλαδή υπάρχει αυτός ο εκδιασμός όσον αφορά τον αποκλεισμό της Ουκρανικής αγοράς εάν αρχίσει το 2015 η Ουκρανία να υλοποιεί την Συμφωνία Σύνδεση. Αυτό με, με είναι απαράδεκτο. Οπότε θα πρέπει η Ένωση και τα κράτη-μέλη με μια φωνή να συνομιλούν με τη Ρωσία. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι το να έχουμε Γερμανούς τουρίστες που να πηγαίνουν για διακοπές ε, στην ε, Κρυμαία που την έχει προσαρτήσει η Ρωσία και κάποιους που είναι περσόνανον non να τους υποδεχόμαστε με κόκκινα χαλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χθες στο G20 δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν εάν η Ρωσία θα προσκληθεί να συμμετάσχει στη συνάντηση κορυφής του G20 στην Αυστραλία. Ταυτόχρονα δεν σταματά τις απειλές προς όλους τους γειτονές της η Ρωσία. Μόλις λίγες ε, μέρες προηγουμένως πριν είπε ότι θα μπορούσε να κάνει ο Πούτιν μια στατιωτική περίπατο σε όλες τις ε, πρωτεύουσες περιοχές της ε, Βαλτικής θάλασσας και της Ουκρανίας κλπ. Και ο, ο Πίτροπος Ντόλγοφ από τη Ρωσία πήγε στην Λετωνία και είπε να προστατεύσει ε, τη ρωσική, ρωσική μειονότητα της χώρας με κάθε μέσον θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα τα λέω για εκείνους που θεωρούν ότι χρειάζεται η ειδική Επιτροπή υποπτήρες εδώ στην ε, ΑΦΕΤ για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω στο θέμα της αποκέντρωσης της Ουκρανίας, γιατί πρόκειται για μια χώρα με πολλές διαφορετικές ε, καταστάσεις. Ε, έχουμε επίσης ε, έχουμε καθολικούς, υπάρχουν καθολικοί, υπάρχουν ορθόδοξοι, αλλά παρόλα αυτά το επίπεδο αποκέντρωσης αφορά οπωσδήποτε την εθνική κυριαρχία της ε, ε, Ουκρανίας. Ε, είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουν μόνοι τους. Δηλαδή γιατί εμείς εάν ζητήσουμε ή απαιτήσουμε την αποκέντρωση της Ουκρανίας τότε επαναλαμβάνουμε ένα επιχείρημα το οποίο έχει χρησιμοποιήσει η ρωσική προπαγάνδα. Μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας βεβαίως για μια, για μια απόφαση που αφορά την αποκεντρωμένη διοίκηση ή το ειδικό καθεστώς των περιφερειών, αλλά τίποτα παραπάνω. Αυτή η χώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει μόνη της ε, τις αποφάσεις της. Ε, μια και μιλάμε για την Ουκρανία η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την ε, Ρωσία ε, πρέπει να πούμε ότι στην ε, ε, Ρωσία έχει αποκατασταθεί η φήμη ενός τρομακτικού εγκληματία. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια και να μην εκφράσουμε την αντίθεσή μας εδώ στην Ευρώπη όταν ε, ε, βάναυση κομμουνιστές ξαναβρίσκουν την φήμη τους. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η διεθνής πολιτική δεν είναι άσκηση επιχάρτου μεταξύ ειδικών για θέματα αυτά και διεθνούς δικαίου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι πολύ ουσιώδες να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική ισορροπία, στρατηγική λόγη. Για παράδειγμα, με εκπλήσει ότι είμαστε τόσο επιλεκτικοί όσον αφορά το μποϊκό της Ρωσίας. Της Ρωσίας είναι το ίδιο, ε, η ίδια απαγόρευση και εμπάργο που ε, κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείες έναντι της Κούβας. Και δεν ε, είμαι υπέρ του γεροντοκρατικού καθεστώτος του δικτατορικού της Κούβας, αλλά είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει να δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα. Δεύτερον, αυτό που ισχύει στην Ουκρανία είναι το ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας στο Κοσφοπέδιο. Όταν ε, υπονομεύσαμε ε, την τελική πράξη του Ελσίνκη και είχε προειδοποιήσει τότε η Ρωσία ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Να οι συνέπειες. Εγώ ήμουν υπέρ τη συμφωνία σύνδεση παρά το ότι έχω πολλές αφιβολίες, γιατί είναι θεμελιώδε για να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Αλλά με εκπλήσει το ότι έχουμε απόλυτα μονόπλευρη άποψη ενώ χρειάζεται διάλογος χωρίς αποκλεισμού. Και διάλογο σημαίνει να συμμετέχουν διάφορες πλευρές. Και υπάρχει μια πλευρά που δεν δεχόμαστε, που μπορεί να θεωρούμε αιρετική, αλλά είναι τμήμα. Άρα πρέπει να συμμετάσχει στο διάλογο. Πρέπει να ακούμε και αυτή την πλευρά. Να τους βλέπουμε, να τους ακούμε. Αυτούς που είναι τμήμα του διάλογου. Και να μην είμαστε μόνο με τους ε, μεν. Έτσι θα βοηθήσουμε το διάλογο. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του συντρόφου Στρεβίτσιους όταν λέει ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση, παρατήρηση των εκλογών. Βεβαίως, συμφωνώ. Συμφωνώ και η αποστολή μας να είναι ως τον δυνατόν πιο πολυάριθμη για να μπορέσει να συμπεριλάβει όλες ε, τις διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Και κοιτάξτε, αυτό θέτει το άλλο θέμα. Οι αποστολές παρατήρησης εκλογών βεβαίως είναι ενδιαφέρουσες, είναι καλές, είναι πολιτική στήριξη που καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητη. Αλλά είναι απλώς μια περιστασιακή ε, παρουσία. Και καλά, ε, δεν είναι δυνατόν ε, να πάμε μόνο σε μερικά εκλογικά, εκλογικά τμήματα και να θεωρήσουμε ότι τα καταλάβαμε όλα γιατί άλλο γίνεται στο Κίεβο, άλλο γίνεται στην Οδυσσό, άλλο γίνεται στη Μαριούπολη. Είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Αυτή λοιπόν η αποστολή εκλογικής παρατήρησης είναι θεμελιώδης. Απόλυτα αναγκαία. Και αυτό που είναι επίσης θεμελιώδε είναι να υπάρχει μία μόνιμη παρατήρηση και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Να ακούμε δηλαδή και την άλλη πλευρά για να καταλαβαίνουμε πλήρως τι συμβαίνει. Άκουσα ορισμένα τύμπανα πολέμου εδώ πέρα. Βεβαίω, εγώ δεν ε, είμαι κατά του να είμαστε στιβαροί όταν χρειάζεται. Όταν υπάρχει για παράδειγμα ε, επιθετικότητα θα δείτε για το Ιράκ ότι θα πω να βοηθήσουμε επιτόπου και να προστατεύσουμε στρατιωτικά τις μειονότητες. Με αυτό συμφωνώ, ήταν δική μου πρόταση. Αλλά τώρα, αυτά τα τύμπανα του πολέμου, η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όταν παράλληλα λέγεται το πρόβλημα είναι η Ρωσία, στρατιωτικά είναι παράλογο. Στρατηγικά είναι ανόητο και το αποτέλεσμα δεν ξέρω ποιο θα είναι. Άκουσα επίσης ότι η Ρωσία προτίθεται να επεκταθεί πέρα από την Μαριούπολη για να υπάρχει χερσαία σύνδεση με την Κρυμαία. Καλά. Αν ρίξετε μια ματιά στο τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γερμανικός στρατός είχε προγεφύρωμα στο Κουμπάν μέσα από τα στενά του Κέρσου για να ελέγχει και τα στενά του Περεκόπ που συνδέουν την Κρυμαία με την Ουκρανία. Να πούμε τώρα ότι τώρα που έρχεται το χειμώνα θα επιτεθούν οι Ρώσοι για να υπάρξει χερσαία επαφή νομίζω ότι είναι ε, ιδιαίτερα απίθανο. Θεωρούμε σίγουρο ότι θα επεκταθεί ο πόλεμος. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό συμφωνεί με την ιστορική πραγματικότητα. Και δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Όχι, να μην υπάρξει περισσότερο πολεμοχαρής προσέγγιση αρκετά πολεμοχαρίσιμα θα μέχρι τώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει διάλογο χωρί εξοπλισμού. Αυτά που είπε ο προηγούμενο ηγητή για την Ουκρανία είναι απόλυτα σωστά. Και αυτά που είπε και ο σύντροφο ο Στρεβίτσιου ω προστίκη και αυτά είναι νομίζω πολύ σωστά. Οπότε, βεβαίω πρέπει να σεβαστούμε την εδαφική ακαιρεότητα τη Ουκρανία και με βάση και την κοινή λογική που προκύπτουν από τη γνώση των στρατηγικών ε, γεγονότων τα καταλαβαίνουμε απόλυτα όταν μας αφορούν. Ενώ είμαστε πολύ εμπλεκτικοί όταν ε, ε, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις άλλων. Παρακαλώ, κοινή λογική, όχι ακαδημαϊκή προσέγγιση καθηγητών διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά έχουν υποθεί ήδη. Εγώ ένα πράγμα θέλω να αναφέρω εξεπλάγην γιατί στη διάσκεψη των Προέδρων ενεκρίθη επταμελής αποστολή για την παρατήρηση των εκλογών στην Ουκρανία. Εξεπλάγην διότι στην ομάδα που ασχολείται με τις εκλογές οι πολιτικές ομάδες είχαν όλες συμφωνήσει η αντιπροσωπεία να είναι πολυπληθέστερη και εξεπλάγην επίσης γιατί πριν από τρία χρόνια όταν έγιναν οι πρώτες εκλογές στην Τινησία είχαμε στείλει 15 μελή αποστολή και ο Μιχαήλ Γκάλερ μου θύμισε ότι στην Παλαιστίνη στις εκλογές είχαμε στείλει 30 μέλη. Επομένως ε, τα συμπεράσματα είναι εύκολα. Δηλαδή τα γράφουμε, τη γράφουμε την Ουκρανία στα παλιά μας τα παπούτσια και συγγνώμη για την έκφραση λέει ο μιλητής θέλουμε να κάνει η χώρα αυτή μεταρρυθμίσεις. Μιλάμε για μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα ε, και ε, όταν φτάνουμε στις εκλογές και μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο είναι η παρατήρηση των εκλογών, ε, στέλνουμε 7 ανθρώπους. Τι θα κάνουν αυτοί οι 7 άνθρωποι επί τόπου. Αυτό είναι το μήνυμά μου και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα ε, χειροκροτήματα αυτών που δεν άκουσαν ότι έχουμε ήδη αποφασίσει να στείλουμε μια επιστολή να ζητήσουμε περισσότερα μέλη να πάνε σε αυτή την αντιπροσωπεία. Με συγχωρείτε που τα λέω τώρα. Ο κύριος Γκάλερτ. Α, με, με, Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Να ακούστε και το εξή. Υπάρχει αυτή η πρόταση γίνεται ε, με βάση τις ε, αυτόματες διαδικασίες της διοίκησης και μπορεί να αλλάξει μόνο με απόφαση του Προεδρείου. Άρα οι συντονιστές μπορούν να συζητήσουν με τους Προέδρους των ομάδων τους, με τον Γενικό Γραμματέα, ούτω ώστε η διάσκεψη των Προέδρων να λάβει άλλη απόφαση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Θα στείλω μια επιστολή, αλλά θα έχει αποτέλεσμα μόνο αν έχετε μιλήσει με τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων για να αλλάξει απόφαση το Προεδρείο. Αυτή είναι η διαδικασία. Η διαδικασία γίνεται από τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να τους ε, ενημερώσετε για να αλλάξουμε την απόφαση. Μήπως αυτές τις επιστολές θα μπορούσαμε να τις στέλνουμε επίσης και στους συντονιστές, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να ξέρουν ότι πρέπει να ενημερώσουν τους ε, προέδρους ε, των ομάδων τους αυτομάτως να κοινοποιούνται στους συντονιστές. Και παρακαλώ επίσης οι συντονιστές να ε, παίρνουν μετά το λόγο. Κύριος Τέρνερ, εγώ ο κύριος Τάνοκ, εγώ θυμάμαι και την επανάσταση, την πορτοκαλιά επανάσταση το 2004 και η αντίστροφη διαδικασία είχε ακολουθηθεί. Οι πολιτικές ομάδες στέλνουν αντιπροσωπείες οι οποίες εγκρίνονται από την εκλογική επιτροπή στην Ουκρανία. Ε, είχαμε στείλει πολλού στην Ουκρανία το 2004, άλλοι από τις πολιτικές ομάδες, άλλοι από το Κοινοβούλιο και είχαν ισότιμο καθεστώ παρατηρητού των εκλογών. Θα πρότεινα λοιπόν μερικές από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες να στείλουν δικές τους αντιπροσωπείες να προσθεθούν στην αντιπροσωπεία τη Επιτροπή. Πρόεδρο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για τι εκλογέ τι ίδιε. Γιατί πόσοι ακριβώ παρατηρητέ θα είναι. όπως είπα, πρέπει και πριν τι εκλογέ να πάμε και στην Οδυσσό και άλλοι όχι μόνο στο Κίεβο. Τι έννοια έχει να πάνε όλοι στο Κίεβο. Να πάνε οι αντιπροσωπείες μόνο στο Κίεβο και τα μεμονωμένα μέλη να πάνε στην ε, ε, επαρχία. Να δείξουμε την παρουσία μας και στην Οδυσσό και σε άλλα μέρη τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Αυτό μπορούν να το οργανώσουν μόνο οι πολιτικές ομάδες, όχι το Κοινοβούλιο. Και καλό λοιπόν τις πολιτικές ομάδες να το κάνουν. Για αυτό το θέμα. Επίσης, εάν δεχθούμε την παρέμβαση της ε, απόφασης, αυτό θα δημιουργήσει προηγούμενο και θα γίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις. Άρα θα πρέπει τα δύο αυτά ζητήματα να μείνουν τα Καλά, λέει ο Πρόεδρος. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά από λίγες εβδομάδες αν έχουμε κάποια παρόμοια ανάγκη. Συμφωνείτε, κύριε Γκάλα. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω. Γιατί το ανέφερε ένας συνάδελφος. Ο αριθμός που θα στείλουμε εμείς ως κοινοβούλιο δείχνει τι πολιτική σημασία αποδίδουμε στις εκλογές. Η μακροπρόθεσμη παρατήρηση της κατάστασης στην Ουκρανία θα γίνει από τον ΟΑΣΕ. Αυτό θα γίνει και ενώπιση των εκλογών αλλά και πριν και μετά και κατά τη μέρα των εκλογών για να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες. Η παρουσία μας είναι πολιτική. Και αν πούμε ότι θα στείλουμε 7, δείχνουμε ότι είναι ως οποιασδήποτε εκλογές αυτές οι εκλογές. Πιστεύω ότι πρέπει τουλάχιστον να διπλασιάσουμε, να πάμε 15, όπως την προηγούμενη φορά. Τώρα για τις ίδιες εκλογές. Με απογοητεύει κάπως το ότι δεν κατέστη δυνατόν, δεν υπήρξε πλειοψηφία, να αλλάξει ο εκλογικό νόμο πριν τι εκλογέ. Άρα θα εφαρμοστεί το προηγούμενο εκλογικό σύστημα. Οπότε, δυστυχώ, η κατάσταση θα είναι σε μεγάλο βαθμό μία από τα ίδια. Και για τι εκλογικέ περιφέρειες υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι κατεβαίνουν ως ε, ανεξάρτητοι, οι οποίοι είναι τσιράκια των ε, ολιγαρχών. Θα προτιμούσα ένα πιο αναλογικό σύστημα και ένα ε, ελάχιστο όριο 5%. Υπήρχε ε, για το θέμα αυτό, υπήρξαν συστάσεις και της Επιτροπής της Βενετίας. Αλλά αυτό που κάνουν τα κόμματα εκεί είναι ότι στα ψηφοδέλτια τους βάζουν εκπροσώπους και από την Κρυμαία και από τον Ντανιέτς και από τον Λουγκάνσκ οπότε θα υπάρχουν εκπρόσωποι από αυτές τις περιοχές στο Κοινοβούλιο Κατά τα άλλα, μία ερώτηση στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης για την παρουσία του ΟΑΣΕ. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο τα κράτη-μέλη μας να μην στέλνουν αρκετά άτομα ούτω ώστε να μπορεί να κάνει ε, τη δουλειά του ο ΟΑΣΕ. Μίλησα με τον Ελβετό πρέσβη στο Κίεβο και μου είπε χρειαζόμαστε πεπειραμένους αξιωματικούς που να μπορούν να κρίνουν τι γίνεται, πώς έχει πολιτικά η κατάσταση. Τους χρειαζόμαστε. Και οπότε αναρωτιέμαι, μα μπορούμε να αποσπάσουμε αξιωματικούς και έχουμε έμπειρους αξιωματικούς. Γιατί λοιπόν αργούν τόσο πολύ <coughs> τα κράτη-μέλη μας καθυστερούν στην ενδυνάμωση αυτής της αποστολής του ΟΑΣΕ. Θεωρώ ότι πολιτικά είναι απαράδεκτο και σημαντικό επίσης να μην παρατηρούμε μόνο τα σύνορα κάνοντας ε, περιπολίες μέσω του ΟΑΣΕ, αλλά και στα κατεχόμενα εδάφη να παρατηρούμε πώς δρούν οι διάφορες ομάδες, αν έχουν δώσει ρωσικά διαβατήρια, αν τους έχουν μοιράσει ρωσικά ε, διδακτικά βιβλία, εάν λοιπόν προωθούν την προσπάθεια προσάρτησης στη Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει επίσης διαφάνεια στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Θα πρέπει να είναι παρόν και ένας Ρώσος εκπρόσωπος και κατόπιν πρέπει να δημοσιεύονται αυτά που είδαν από κοινού. Μόνο έτσι μπορεί να αυξηθεί η πίεση στη ρωσική πλευρά να είναι πιο επιφυλακτική, να σταματήσει να δημιουργεί επιτόπου de facto κατάσταση προσάρτησης όπως και στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο. Α. Ιράκ ακούμε τις τελευταίες λέξεις του Πρόεδρου. Και αυτό είναι κρίμα. Οπότε Θα δούμε πώς θα το επιτύχουμε. Είναι δυνατόν μήπως ε, σήμερα το απόγευμα. Μάλλον εννοεί τη συζήτηση για τα θέματα Ιράκ Συρίας. Γιατί ξέρετε έχουμε και αυτά τα άθλια πράγματα με την οποία ελέγχουν του προπολογισμού. Ε, ναι, μας είπαν να πάμε στην αίθουσά τους γιατί αυτή είναι η αρμόδια επιτροπή και άλλα τέτοια. Έχετε καμιά πρόταση πώς μπορεί να γίνει αυτό. Παρουσίαση. Νομίζω. Όχι, όχι την επόμενη συνεδρίαση. Είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό όπως ε, ένα κατεπήγον θέμα όπως η Ουκρανία. Σας παρακαλώ, Η επόμενη ένα λεπτό ο καθένας. Ένα λεπτό ο καθένας, σαν επεξηγήσει ψήφου. Στετίνα ο επόμενος. Και μετά η κυρία Λόζινγκ. Ένα λεπτό έκαστος. Ευχαριστώ. Εγκρίνω την πρόταση να στείλουμε περισσότερους στην Ουκρανία ευρωβουλευτές και προτείνω να μην σταλούν μόνο ε, στις περιοχές που αναφέρατε, θα πρότεινα οι συνάδελφοί μας να πάνε και στην περιοχή του Ντανιέτσκ στο Σλαβιάνσκ για παράδειγμα, στο Κραματόρσκ και στο Αρτεμόσκ. σε όλες αυτές τις περιοχές είναι πολύ σημαντικό διότι πιστεύω ότι θα είχε μεγάλη συμβολική αξία Τώρα από πλευρά ε, πρακτική δυνατότητα είναι δυνατόν. Η κατάσταση είναι σχετικά ασφαλή σε αυτέ τι περιοχέ τώρα. Και νομίζω ότι οπωσδήποτε θα έχει μεγάλη δημοσιότητα μια τέτοια παρουσία μα, θα δείξει πόσο στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις περιοχές αυτές. Το λέω από τη δική μου την πείρα. Πρόσφατα ήμουν σε αυτές ε, τις περιοχέ, και ξέρω με πόση χαρά με υποδέχτηκαν ω απλό Ευρωβουλευτή και πώς με καλωσόρισαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Ευχαριστώ. Η επόμενη. Η κυρία Λόιζεν. Νομίζω ότι υπήρξαν διαφορετικές απόψει των συναδέλφων. Ορισμένοι στην ουσία υποδαβλίζουν την ένταση με αυτά που λένε κατά τη γνώμη μου. Άλλοι έχουν μια πολύ, μια, μια πολύ πιο μετριοπαθή στάση. Αναφέρθηκε ήδη η στάση μας για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Χαίρομαι πολύ που το εμπορικό τμήμα της συμφωνίας έχει παγώσει προς στιγμή διότι προσπαθούμε να υπάρξει μια ερνευτική διαδικασία, να ξεκινήσει. Χρησιμοποιήθηκε ο όρος ε, οικονομική κατάπαυση του πυρός. Στηρίζω αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό σημαίνει ότι προηγουμένως υπήρχε εμπορικός πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Άρα και η συμφωνία αυτή είναι όπλο δεν είναι απλώς ένα οικονομικό θέμα. Υπάρχει και οικονομικός πόλεμος. Προτείνω λοιπόν να ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να απόσχουμε από στάσεις που ακούστηκαν και εδώ ότι δεν θα πρέπει καθόλου πλέον να διαπραγματευόμεθα με τη Ρωσία. Η Ουκρανία είναι μια χώρα όπου υπάρχουν βαθιές διαφορές και μετά τις εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό η στάση μας να βοηθήσει τη διαδικασία ειρήνης και συμφιλίωσης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Να βοηθήσουμε βεβαίως και διάφορες τομεακές μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτό είναι πιο σημαντικό. Πρόεδρος, ξέρετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ουκρανών στη δημοσκοπήση είναι υπέρ της ενότητας της χώρας και όπως ξέρετε το κοινοβούλιο τους ομόφωνα ψήφισε την επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Ποιες είναι οι διαφορές, ποια είναι τα βαθιά χάσματα. Ε, το χάσμα προκλήθηκε από την ε, ε, ρωσική εισβολή. Βέβαια, οι ιδεολογίε δεν σε επιτρέπουν να το δείτε αυτό, αλλά έτσι έχει η κατάσταση. Κύριο Πέταρ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, λέει ο κύριος Πέτερ, παρά αυτή την κεχηρία που δεν εφαρμόζεται και παρά την ε, ασυμμετρία όσον αφορά την υλοποίηση της σύμφωνας Σύνδεσης, εγώ είμαι αισιόδοξο για το μέλλον και ελπίζω ότι τελικά πρόκειται να στεριώσει η διαδικασία ειρήνευσης. Ε, δεν θέλω να αποτύχουν αυτές οι προσπάθειες. Η δε συμφωνία σύνδεσης μας βοηθάει να επηρεάσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Όμως θα πρέπει να γίνουν και άλλα. Λόγω της πόλωσης πολλά δεν έχουν γίνει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε προς εθνική συμφιλίωση. Και αυτό θα γίνει εάν προχωρήσει προς τα μπρος η χώρα. Χρειάζεται να υπάρχει κάποια συνέχεια, κάποια δυναμική, κάτι το οποίο λείπει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστες οι μεταρρυθμίσεις όπως και το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτή η ομάδα που συγκροτήθηκε είναι κάτι θετικό. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο ε, Οστρεβίτσιους ότι η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε και να προγραμματίσουμε για τον χρόνο μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι την εμπειρία μας μπορούμε να την μεταλαμβαδεύσουμε στην Ουκρανία. Όχι, δεν θέλουμε να παρέμβουμε στα ιστορικά τη ε, Ουκρανία, Αν θέλετε να παρέμβετε, να το πείτε ανοιχτά. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Λέω κύριε Σκέλα. χώρα και έγινε αυτή η κύρωση Οπότε έτσι διάλεξε να ασκήσει το κύριο δικαίωμα, τόσο ώστε να μπει, ε, να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία, στον Ευρωπαϊκό Κράτο Δικαίου. Είναι διχασμένη η χώρα, όχι από το λαό τη, αλλά από τον ξενοπαράγοντα. Και το προβληματικό είναι το ότι αν πασχίσουμε να ζητήσουμε μια πολιτική λύση, ε, τότε θα μπερδέψουμε τα πράγματα. Γιατί η Ρωσία αρνείται ότι έχει εισβάλλει, αρνείται ότι διατηρεί στρατό. Από την άλλη μεριά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι ειδικοί στα στρατιωτικά μας είπαν ότι τα πιο σύγχρονα ρώσικα όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Κάτι το οποίο είναι συγκρίσιμο με τακτικά ε, ατομικά όπλα. Και έτσι εκαθάρισαν, γκρέμισαν, ισοπαίδωσαν ολόκληρα τμήματα πόλεων. Και ξαναγυρίζουμε τώρα στο πιο βασικό. Αυτό είναι μια σύγκρουση αξιών και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Ουκρανίας. Είναι το θέμα εδώ το κατά πόσο θα πρετανεύσουν οι διεθνείς συνθήκες, το διεθνές δίκαιο, το κράτος δικαίου κλπ. Οπότε μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό το κατά πόσον θα πρέπει να κάνουμε κάτι να αξιολογήσουμε το τι έγινε στα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Εάν είχαμε κάνει αυτή την εκαθάριση, αυτή την κρίση που χρειαζόταν, ε, τώρα δεν θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον Πούτιν. I will speak in Spanish, me quiero... Θα μιλήσω στα Ισπανικά γιατί Βοηθώ στους συναδέλφους που συνέγκριναν το Κόσοβο με την ε, Κρυμαία και επειδή εδώ πέρα έχουμε ασχοληθεί με το Κόσοβο, σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τέτοιου σύγκριση και καμία κυβέρνηση στο Κίεβο έκανε αυτά τα οποία έκανε το ομιλόσεβιτ του Αλβάνο Κοσοβάρους. Και από πλευρά διοίκηση, από πλευρά πολιτική τι έγινε τόσα χρόνια και κατόπιν εξαπέλυσε και πόλεμο και σκότωσε τόσο κόσμο και από την άλλη μεριά. Το Διεθνές Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2010 είπε ότι με την ε, διακήρυξη της Βενετίας δεν είχαμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Οπότε παρακαλώ, πέραν των θεμάτων των Ισπανικών, ε, να μην συγκρίνετε την Κρυμαία με το κρυσφοπέδιο als Berichterstatter in einer Ο κύριος Αρσβόλσκι είναι εισηγητής, δεν ξέρω. Εσείς αν θα μπορείτε να μας συνοψίσετε όλη τη συζήτηση, αν έχετε κάποιο είδου ε, πρόταση που να φέρει συνένεση. Σάρις Σε ευχαριστώ, Χέλμαρ. Εδώ είναι πόλεμος και εμείς μιλάμε για ε, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες. Η, Ρου... Ρωσία θέλει απλώς την Ουκρανία, ολόκληρη την Ουκρανία, τη θέλει πίσω, τη θέλει δικιά της. Δεν υπάρχει πάυση πυρός στην ουσία και αναρωτιέμαι τι θα συζητήσουν στην Κορεπέρ οι ε, πρέσβεις, την, το να γίνουν οι ποιότερες ε, οι, ε, οι κυρώσεις. Το αντίθετο θα έπρεπε να γίνει. Και νομίζω ότι θα πρέπει από τη στιγμή που υπάρχει περισσότερος πόλεμος να υπάρχουν και περισσότερες κυρώσεις. Και βεβαίως σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία. Και όλα τα αξιόπιστα στοιχεία, πέρα από τα ψέματα που λέει η Ρωσία, που λέει ότι δεν θέλει να παρέμβει και τα λοιπά. Εάν τα πιστέψουμε αυτά, τότε ε, θα βρεθούμε κάποια στιγμή ε, ε, ενώπιον προ, εκπλήξεων, γιατί όπως λέει και ο πρόεδρος Μπροκ, θα ανοίξει πρώτα ένας χερσαίος διάδρομος και μετά θα φτάσουμε στην υπερνηστερία και μετά στο δέλτα του Δούναβη και κλπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Είτε θα αποσταθεροποιήσουμε τη Ρωσία με περισσότερες κυρώσεις πριν πάρει τα πάνω της και προχωρήσει περισσότερο ή διαφορετικά θα κάνουμε όλο και λιγότερα και τελικά θα χαθούμε και εμείς, θα, χάσουμε και την, θα χαθεί και η Ουκρανία και θα προχωρήσουμε σε καταστάσεις ε, οι οποίες ε, ε, θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να αναλυφθούν, δηλαδή να σταματήσουμε ε, να, να πουλάμε όπλα στην Ουκρανία, θα πρέπει να βγάλουμε την Ρωσία από την Ατομική Συμφωνία. Ε, εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι μετά από απόφαση του Συμβουλίου έπρεπε να αρχίσουμε να πουλάμε ξανά όπλα στην Ουκρανία. Αλλά επειδή φοβόμαστε έχουμε σταματήσει την πώληση των όπλων. Ναι, δεν ήταν ακριβώς αυτή η συμφιλίωση που ε, θεωρούσα εγώ ότι πρέπει να ισχύσει. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια δυνατότητα να συντομεύσουμε την ακρόαση με τον εκπρόσωπό μας στην ε, Ιαπωνία και να πάμε ένα τέταρτο αργότερα στην ακρόαση με την Επιτροπή Κόντ και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μισή ώρα για την συζήτηση για Ιράκ και Συρία. Ποιο συμφωνεί? Υπάρχει κανεί που να διαφωνεί? Α, εσείς βλέπω ότι συμφωνείτε ο κύριε Πάσχου, οπότε θα σας δώσω και την Προεδρία για τη συνάχεια. Λοιπόν, προτείνω τώρα 35 λεπτά για την Ιαπωνία. Τώρα είναι θέμα δικό σας να είστε σύντομοι σε ερωτήσεις σας. Ε, δεν πρόσεξα από την αρχή το χρόνο μιλίας που έδινα. Ορισμένοι μίλησαν 10 λεπτά και μετά γύρω στις 11 και 10 να αρχίσει η συζήτηση για το Ιράκ και τη Συρία και 12 παρατέταρτο να πάμε στην άλλη επιτροπή. Εδώ δύο ορόφους παραπάνω. Συμφωνείτε? Παρακαλώ, ε, μπορείς να αναλάβεις την Προεδρία.